Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Κυρίες και κύριοι, καθίστε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Ήδη έχουν περάσει τέσσερα λεπτά μετά τις τρεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με την σημερινή και αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής ΙΝΤΑ, Διεθνούς Εμπορίου. Το πρώτο σημείο της σημερινής διάταξης είναι η έγκρισή της. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν αν έχετε κάποιες αντιρρήσεις, δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη ως έχει. Σημείο 2. Πρακτικά, έγκριση των πρακτικών. Η συνήθις διαδικασία είναι ότι μέχρι το τέλος αυτής της συνεδρίασης θα πρέπει να υποβάλλετε αντιρρήσεις και σχόλια, εάν υπάρχουν. Αλλιώς εγκρίνονται τα πρακτικά ως έχουν. Και αυτό ακριβώς θα ακολουθήσουμε σαν διαδικασία και αυτή τη φορά. Και περνάω στο σημείο 3. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο οι διάφορες πληροφορίες για τις συνεδριάσεις στο Τάλιν, στη Ρώμη, στη Λισαβόνα, στο Λίνεμπορκ και φυσικά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ήδη έχουν ενημερωθεί. Πιστεύω ότι όσοι δεν το έχουν κάνει πρέπει να το κάνουν ε, άμεσα. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι όσον αφορά τις πολύ πρόσφατες διαπραγματεύσεις, η συμφωνία εδώ στο Κοινοβούλιο για καλύτερη νομοθεσία καθώς και η διοργανική συμφωνία που βεβαίως μας αφορά, καθώς και ο τριμερής διάλογος και η συνάντηση που θα λάβει η χώρα. Κυρίως όμως εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρέπει να προσέξουμε είναι οι διαπραγματεύσεις με τους ε, δύο άλλους θεσμούς, η βελτιωμένη δηλαδή συνεργασία όσον αφορά τις ε, εξωτερικές σχέσεις, την εξωτερική πολιτική Ξέρετε ότι η διοργανική συμφωνία έχει επεξεργαστεί όλες αυτές τις πτυχές, καθώς και τη δική μας συμμετοχή και σύμφωνα με την συμφωνία αυτή και την, τον 12ο γύρο συνομιλιών. Οι υπεύθυνοι για τελωνιακά θέματα δείχνουν ε, από τα συμπεράσματά τους ότι σαφώς ε, στα πλαίσια του ΠΟΕ προχωράνε οι διαπραγματεύσεις και ότι τα πολύ πρόσφατα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Στις 17 Μαρτίου από την κοινή διαβούλευση για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με την Κίνα καθώς και την συνδιάσκεψη TDI και βεβαίως εγώ θα είμαι παρόν, θα γίνουν και τα εισαγωγικά σχόλια. Έχουμε, όπως ξέρετε, τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι σαφώς και θα εκφράσουν τις γνωστές θέσεις της Επιτροπής. Τώρα, θα περάσω στο σημείο 4 αμέσως. Έχουμε έναν παλιό μας γνωστό, τον Jean-Luc Marti από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζων θα συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων και τα 30 πρώτα λεπτά, η πρώτη μισή ώρα, θα αφιερωθεί στην συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, δηλαδή την συμφωνία ΣΕΤΑ. Φαντάζομαι ότι θυμάστε ότι στις 29 Φεβρουαρίου ο, η υπουργό ε, αρμόδια του Καναδά για τις εμπορικές σχέσεις καθώς και η Σεσίλια Μάλστρομ φυσικά στα πλαίσια του νομικού σουέμπινγκ συναντήθηκαν οδήγησαν στο καινούργιο κείμενο, το οποίο βεβαίως ε, είναι ως ένα σημείο ανανεωμένο με κάποιες ε, συγκεκριμένες ε, αλλαγές, τροποποιήσεις. Το νέο κείμενο έχει μεταφραστεί, μεταφράζεται μάλλον αυτές τις μέρες και φυσικά θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την τελική υπογραφή. Έχουμε κάποιο χρόνο μέχρι την ημερομηνία της τελικής υπογραφής για να μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε περαιτέρω και να δούμε τις μικρές αλλαγές. Ο Σον Λουίκ Δεμαρτή θα μας κάνει μια πρώτη παρουσίαση για το τελικό κείμενο της συμφωνίας όπως το γνωρίζουμε. Κατόπιν φυσικά θα δώσω το λόγο και στον εισηγητή, στους Κιώδης και σε όποιον άλλο θέλει να πάρει το λόγο. Καταρχήν δίνω το λόγο στον Ζων Λουίκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Μπέρντ. Αξιότιμα μέλη, έχουμε καλά νέα για τη ΣΕΤΑ. Δεν ξέρω αν επειδή είναι καλά τα νέα είναι λιγότεροι στην αίθουσα. Εν πάση περιπτώσει, η νομική αναθεώρηση του κειμένου έχει ολοκληρωθεί και τώρα έχουμε ένα πραγματικά τελικό κείμενο. Το αναθεωρημένο κείμενο περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις στο κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Πέρα από την ενδελεχή συζήτηση που έγινε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αξιωματούχους του Καναδά, είχαμε την ολοκλήρωση όλων αυτών των συζητήσεων μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα κυβέρνηση του Justin Trudeau και το πλήρες κείμενο από τη ε, Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Η νέα προσέγγιση που ε, συμφωνήσαμε τους Καναδούς και που στηρίζει η νέα Υπουργό Εμπορίου κυρία Φρίλαντ θεσπίζει ένα σύστημα πιο δίκαιο, πιο σόφρον, πιο διαφανές έχουμε πλήρη διαφάνεια των διαδικασιών. Ξεκάθαρα πρότυπα προστασίας για τους επενδυτές, για παράδειγμα για τις έμεσες απαλωτριώσεις, δεν υπάρχει αμφισμία ούτε υπερβολικές διεκδικήσεις, πράγματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Τα κράτη έχουν το δικαίωμα να νομοθετούν βεβαίως προς το συμφέρον του ε, το δημόσιο. Υπάρχει κώδικας δεοντολογίας για την ανεξαρτησία των διαιτητών στη διαιτησία και πολλές άλλες σημαντικές καινοτομίες περιλαμβάνονται. Η ΣΥΤΑ περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της νέας προσέγγισης για την προστασία των επενδυτών και για την επίλυση των ε, διαφορών, όπως το ζήτησε άλλωστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας παραθέτω τα εξής. Ένα νέο άρθρο που διατηρεί το δικαίωμα του νομοθετήν για θέματα δημόσιας πολιτικής σε όλα τα επίπεδα ε, κυβέρνησης, διακυβέρνησης και διοίκησης. Δεύτερον, δεν θα υπάρξει ad hoc διαιτησία. Δεν θα υπάρξει πια αυτό στη ΣΥΤΑ. Θα υπάρξει ένα δικαστήριο μόνιμο, θεσμικό, θεσμοθετημένο, για την επίλυση των διαφόρων και τα μέλη του δικαστηρίου δεν θα οριστούν από τους επενδυτές και από τα κυρίαρχα μέρη, από τους επενδυτές, αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Καναδά. Θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα προσόντα και θα έχουν τυχαία επιλογή και ανάθεση υποθέσεων και φακέλων, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αμεροληψία και να μην υπάρχει αμφιβολία για την αμεροληψία τους. Και θα, υπάρχουν, θα υπάρχει και επιτροπή δολοντολογίας για να εντοπίζει τις συγκρούσεις συμφερόντων. Δεν μπορεί κανείς να έχει δύο ιδιότητες. Δεν μπορεί να δουλεύει ως δικηγόρος ή νομικός εμπειρογνώμονος σε οποιαδήποτε άλλη επίλυση διαφοράς για θέματα επενδύσεων όταν είναι μέλος του δικαστηρίου αυτού και ε, διαιτητεύει για συγκεκριμένη υπόθεση. Όλα αυτά είναι συγκρίσιμα με αυτά που υπάρχουν στις ε, χώριες ένομες τάξεις. Και έχουμε συγκεκριμένες προβλέψεις για τη διοντολογία, για το, τους λόγους για τους οποίους μπορεί κανείς να ασκήσει έφεση, αλλά και για τα προσόντα. Και η αμοιβή θα προσαρμοστεί γρήγορα από την Σχετική Επιτροπή για την παρακολούθηση της θέσης σε ισχύ της ΣΥΤΑ, της Συμφωνίας ε, Εμπορίου και Επενδύσεων με τον Καναδά. Ορισμένοι έχουν θεωρήσει ότι η προσέγγιση αυτή είναι κάπως μη δημοκρατική και θεσπίζει ένα παράλληλο σύστημα που ε, δεν θα περάσει τη δοκιμασία της πολιτικής και δημοκρατικής νομιμοποίησης. Όμως, η νέα Καναδέζικη κυβέρνηση και εμείς απορρίπτουμε αυτό το σκεπτικό, διότι το νέο ε, σύστημα ε, δικαστηρίων επίλυσης επενδυτικών διαφορών στηρίζεται πλήρως από ε, εκλεγμένες κυβερνήσεις και κοινοβούλια. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα για την επενδυτική μας πολιτική και δείχνει τη σοβαρότητά μας κατά την ε, εφαρμογή αυτής της ε, πολιτικής. Υπάρχει και η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου η νέα Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου η οποία θα ενισχύσει την επενδυτική μας πολιτική. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το εγχείρημα. Βλέπουμε ότι και άλλοι εταίροι την ε, υιοθετούν. Γιατί λοιπόν η ΣΥΤΑ είναι μια καλή συμφωνία. Διότι είναι μακράν η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με το μεγαλύτερο ευελινικές που έχει επιτευχθεί ποτέ σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά. Θέτει νέα πρότυπα για τους κανόνες για τις επενδύσεις και αυτό είναι σημαντικό μήνυμα και στους άλλους εταίρους με τους οποίους έχουμε εμπορικές σχέσεις. Δείχνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει συνολικές και φιλόδοξε συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου με, τους βασι... με τι βασικές χώρες τις οποίες εξάγει ή οι οποίε εξάγουν σε αυτήν εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέτοντας νέα πρότυπα. Έχουμε νέα πρόσβαση στην αγορά, πολύ καλύτερη και σε τομείς που είναι που ενδιαφέρουν πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσπίζεται νομική ασφάλεια, νομική βεβαιότητα σε πάρα πολλούς τομείς. Ε, υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα για τους παρόχους υπηρεσιών, διευκολύνει η συμφωνία την μεταφορά βασικού προσωπικού από τη μία μεριά του Ατλαντικού στην άλλη, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ε, προσλαμβάνουν για after-sale services, για διάφορα προϊόντα και για διάφορους τομείς, και θα δημιουργήσει το πλαίσιο για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε τομείς που είναι ρυθμισμένοι από τα κράτη όπως είναι ο κλάδος των αρχιτεκτώνων ή των λογιστών, των ορκωτών ελεκτών και το καθεξής. Και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να νομοθετούν όταν πρόκειται για δημόσια υπηρεσία με τον τρόπο με τον οποίο θεωρούν το πιο κατάλληλο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για να αναλάβουν την πώληση αγαθών, την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης στον Καναδά, σε επίπεδο επαρχίας, δήμων ή κεντρικής κυβέρνησης. Δίνεται πρόσβαση στην αγορά στα γαλακτοκομικά και για τα μεταποιημένα προϊόντα καταργούνται οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και οι δασμοί. Είναι η πρώτη συμφωνία με μια χώρα η οποία παραδοσιακά ήταν εξαιρετικά επιφυλακτική με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Θα προστατεύσει ο Καναδάς 145 γεωγραφικές ενδείξεις με ένα σύστημα που μοιάζει με το δικό μας. Ε, με αυτή την συμφωνία θα υπάρχει μεγάλη ε, εξοικονόμηση στις εξαγωγές αγαθών όταν έχουμε να κάνουμε με το double tasting. Δεν θα χρειαστεί διπλή πιστοποίηση για, σε διάφορους τομείς όπως είναι οι οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές, ε, ηλεκτρονικές συσκευές, μηχανήματα και κ.ο.κ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τον Ιούνιο τον αργότερο το Σώμα των Επιτρόπων να εγκρίνει αυτό και να το υποβάλει στη συνέχεια ε, στο Συμβούλιο διαβουλευόμενη Επιτροπή με το Ευρωκοινοβούλιο ταυτόχρονα θέλουμε να υπογραφεί μαζί με το SPA, τη Συμφωνία για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση, τον Οκτώβριο και στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο για τη συγκατάθεσή του. Είναι μια εμπορική συμφωνία καινοτόμος που ε, θεσπίζει νέους κανόνες για τις επενδύσεις και ανοίγει ε, την πρόσβαση σε αγορές. Έχουμε ε, προσέξει ιδιαίτερο και ε, λάβει υπόψη μας το μέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι όπως ε, το τονίσατε στις εκθέσεις που εγκρίνατε στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Δεν ήταν εύκολο αυτό το εγχείρημα. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε πλήρη συνείδηση του πόσο σημαντικό είναι αυτό το καθήκον που έχουμε αναλάβει. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι έχουμε αφουκραστεί τις ανάγκες και τα αιτήματά σας και τα έχουμε πλήρως λάβει υπόψη. Η νέα κυβέρνηση του Καναδά έκανε και αυτή πολύ σημαντικά βήματα απομακρυνόμενη από το υφιστάμενο σύστημα και η πλευρά αυτή δεν επιθυμεί περαιτέρω αλλαγές στην συμφωνία. Η νέα κυβέρνηση του Καναδά προσυπογράφει πλήρως αυτή την προσέγγιση, την επιθυμεί. Με αυτή τη συμφωνία θα έχουμε υψηλότερα πρότυπα και αυτά είναι καλά νέα για τους καταναλωτές, για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις μας. Ελπίζω να είμαστε σε θέση να αγγιθούμε στους πολίτες μας και στις επιχειρήσεις μας, τις μικρομεσαίες και τις μεγάλες, ότι θα επικυρωθεί αυτή η συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Και σας ευχαριστώ για τη στήριξη και τη συμμετοχή σας. Τέλος, είναι σαφές ότι τέτοιου είδους συμφωνίες δεν αποσκοπούν στο να υπάρξει μια πλήρως ενιαία αγορά ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Δεν ήταν αυτός ο στόχος, ούτε πρόκειται να συμβεί αυτό ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ τον Ζολίκ για αυτή την εισήγηση για τη Συμφωνία ΣΥΤΑ. Νομίζω ότι υπάρχουν οκτώ ομιλητές και έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Περισσότερο ως προς τη διαδικασία δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες τώρα και σίγουρα θα έχουμε και τη διαδικασία κύρωσης μπροστά μας. Έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας δηλαδή για να συζητήσουμε τη Συμφωνία ΣΥΤΑ λεπτομερώς. Γι' αυτό θα ήθελα να αρκεστείτε στα δύο λεπτά. Ο κύριος Πάπλεξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για την επιτυχή αναθεώρηση της Συμφωνίας ΣΥΤΑ και νομίζω ότι μπορούμε να συγχαρούμε τους διαπραγματευτές της Επιτροπής. Δηλαδή, ανταποκριθήκατε στην εντολή του Κοινοβουλίου και καταφέρετε να έχετε και μία αποδοτική πορεία, ένα αποδοτικό αποτέλεσμα σε σχέση με τα, το Διεθνές Δικαστήριο από πλευράς ε, Καναδά. Η ζωή συνεχίζεται και σε αυτό το στάδιο μπορούμε να πούμε με κάθε αξιοπρέπεια ότι η Συμφωνία ΣΥΤΑ κινείται πολύ μακριά και υπάρχει μια ποιοτική συμφωνία. Πολύ πιο ποιοτική από αυτή που αρχικά είχαμε κατά νου. Να σας συγχαρώ λοιπόν και θα ήθελα επίσης να πω ότι από τη δική μου πλευρά ε, είμαι πολύ ικανοποιημένος με το κεφάλαιο για το IDS. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία για το εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Καναδά, αλλά αυτό είναι ένα από τα κεφάλαια τα οποία συζητήθηκαν ευρέως και επιτύχαμε. Αναμένουμε λοιπόν το τελικό έγγραφο για τις συζητήσεις μας και όπως είπε και ο Πρόεδρος θα ήθελα να ακολουθήσουμε μία σύντομη οδό γιατί δεν μπορούμε πια να περιμένουμε. Μόιζε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι αυτά που θα αναφέρω, τα αναφέρω με κάθε επιφύλαξη της ε, συζήτησης που θα γίνει στο Κοινοβούλιο και στην ομάδα μου, την ομάδα των ε, σοσιαλιστών. Γιατί θα πρέπει να κοιτάξουμε εκ του σύνεγγι στο κείμενο για να το κατανοήσουμε απόλυτα. Παρόλα αυτά, θα ήταν άδικο να μην αναφέρω ότι αυτή είναι μία μεγάλη νίκη για το Κοινοβούλιο και για την ομάδα μας η οποία πίεσε για να απομακρυνθούμε από το ISTS και νομίζω ότι έγινε μία ε, μετατόπιση δηλαδή σε σχέση με τις επενδυτικές ε, συμφωνίες το πλαίσιο των επενδυτικών συμφωνιών έχει αλλάξει με βάση το νέο ΣΥΤΑ. Και επειδή δεν θέλουμε να περιαυτολογούμε, θα θέλαμε να συγχαρούμε την Επιτροπή για αυτή την εργασία και αυτό το ποιοτικό άλμα που έγινε για την τροποποίηση της συνθήκης. Αυτό βεβαίως με την επιφύλαξη των μελλοντικών συζητήσεων θα δούμε και θα κρίνουμε το ΣΥΤΑ, τη συμφωνία και δεν θα δούμε μεμονωμένα κεφάλαια ή ένα μεμονωμένο κεφάλαιο, θα κρίνουμε τη συνθήκη στο σύνολό της. Επίσης, θα ήθελα ο Ζαν Λουκ να μας μιλήσει για ορισμένες λεπτομέρειες Θέλετε να σταματήσω. Εντάξει, Πρόεδρε. Πώς ε, βλέπετε αυτό το νέο κατόφλι. Πώς θα επηρεάσει το TTIP. Έμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαστε πολλοί σήμερα, αλλά είναι Δευτέρα Δεν έχει σχέση με εσά ή με το θέμα που συζητάμε. Όσον αφορά την κατάσταση και πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα για το ΣΥΣΑ. Εμείς όσον αφορά τη δικιά μας πολιτική ομάδα, το ECR, φυσικά διαπιστώνουμε ότι γίνονται οι διαπραγματεύσεις και ότι τελικά μας υποβάλλεται ένα αποτέλεσμα όσον αφορά το θέμα των επενδύσεων. Θα ήθελα να ξέρω, θα ισχύσει το πολυμερές σύστημα και πώς θα γίνει αν ε, Πρόκειται για διαφορετικούς εταίρους, ιδιαίτερα όσον αφορά το χρόνο των, διαφόρων επενδύσεων. Βλέπω ότι ισχύει διαφορετική χρονική περίοδος για το TTIP, διαφορετική για την ΣΥΤΑ. Ήδη υπάρχουν πολυμερείς συμφωνίες με τις Ηνωμένε Πολιτείες και στα πλαίσια της Συμφωνίας ΣΥΤΑ πώς θα ρυθμίσετε το θέμα αυτών των πολυμερών ε, διαπραγματεύσεων που αφορούν τις επενδύσεις. Όσον αφορά τώρα τις ε, διαπραγματεύσεις αυτές και τη θέση ισχύ. Μας είχατε δώσει ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του 2016. Αυτό βλέπουμε δεν θα τηρηθεί. Βλέπετε να προχωρεί και στο 2017 η διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι περισσότερες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα για την προστασία των επενδύσεων, έχουν ληφθεί υπόψη. Πρόκειται για διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Καναδά, φιλελεύθερη κυβέρνηση και εμείς πρέπει εδώ να παίξουμε έναν σημαντικό ρόλο και όσον αφορά την προστασία των επενδυτών αλλά και γενικότερα το ε, πλαίσιο αυτών των ε, εμπορικών διαπραγματεύσεων. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε αποστολή στον Καναδά και εγώ θα είμαι μέλος αυτής της αποστολής Πιστεύω θα πρέπει να προετοιμάσουμε σωστά τα επόμενα βήματα αυτή της διαπραγμάτευσης και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί αποφασίσατε να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή από το Κολέγιο των Επιτρόπων μόνο τον Ιούνιο ή μάλιστα τον Ιούλιο από ό,τι κατάλαβα. Χάσαμε πολύ χρόνο και εμείς στην ε, πολιτική μας ομάδα είμαστε πραγματικά διατεθειμένοι και έτοιμοι να προχωρήσουμε ταχύτερα, το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, εγώ δεν είμαι υπέρ του να συνδεθούν ε, οι συμφωνίες TTIP με αυτήν που επεξεργαζόμαστε με τον Καναδά, την ΣΥΤΑ. Ε, από την αρχή ήμουν ε, κατά και πραγματικά πιστεύω ότι κάποια από τα σημεία που θα επεξεργαστούμε στο ΣΥΤΑ μπορούν ενδεχομένως μετά να επεξεργαστούν με τον ίδιο τρόπο και στην TTIP. Ευχαριστώ. Περιμένω να βάλουν όλοι τα ακουστικά τους. Οι 150.000 αν θέλετε αντιρρήσεις δεν έχουν ακόμα απαντηθεί ε, σήμερα διαπιστώνουμε ότι συνεχίζουν να έχουν περισσότερα δικαιώματα και μεγαλύτερη προστασία οι επενδυτές. Σε αυτήν την ε, συμφωνία δεν ε, διαπιστώνω απολύτως καμία πρόοδο και ευχαριστώ την κυρία Ρένα διότι σημείωσε κάποιες από τις αντιρρήσεις μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσετε και αυτά που είπε ο καθηγητής Ντεβίλ και σε καμία περίπτωση να μην ληφθούν προσωρινά μέτρα, ιδιαίτερα για όλους τους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στο Συμφωνία TTIP, Παραδείγματο χάρη πουθενά δεν αναφέρεται η κοινωνική ευθύνη, το θέμα του περιβάλλοντος. Ούτε εκεί βλέπουμε να έχει προχωρήσει η συμφωνία και ούτε στη συμφωνία ΣΥΤΑ ο Καναδάς δεν έχει κυρώσει τις ε, συμβάσεις με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Όλες αυτές οι ανησυχίες σε κάθε περίπτωση παραμένουν και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τεμαρτή, λέει ο κύριος Ζεμπό. Ακούσατε πολλά συγχαρητήρια, αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό Άρμπερ είναι αυτός που καταρχήν θα πρέπει να λάβει τα συγχαρητήριά μας, γιατί πραγματικά προσπάθησε έτσι ώστε 75.000 ε, ε, βόηο κρέας και άλλο τόσο χείριο να μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά και να αποσταθεροποιήσουν ακόμα περισσότερο τους ε, Ευρωπαίους αγρότες Ίσως θα πρέπει εδώ λοιπόν να μην ε, ξεχάσουμε και το θέμα των ε, διαπραγματεύσεων που αφορούν ε, τις το θέμα των ασφαλτοδών άμμων και φυσικά πολλά από αυτά αποφασίστηκαν αντιβαίνουν των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάβασα τις προτάσεις του κυρίου Μπέσσερα για το άνοιγμα των ε, κρατικών προμηθειών και των ε, διαφόρων διαδικασιών και προκηρύξεων διαγωνισμών και διάβασα και τις ε, παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτού του ανοίγματο και πόσο πολύ η Επιτροπή δεν είχε εκτιμήσει ορθά τις επιπτώσεις αυτές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της διευθέτησης των διαφορών, ουσιαστικά αλλάξαμε τίτλο, αλλά στην ουσία παραμένει η ίδια διαδικασία. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις μπορεί να προσφύγουν κατά κρατών. Δεν πρόκειται για δημόσια δικαιοδοτικά όργανα, δεν πρόκειται για δικαστές οι οποίοι υπακούν σε ένα κρατικό δικαστικό σύστημα. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο και πραγματικά εκπλήσωμε γιατί συνεχίζει η δικαιοδοτικο οργανο και πραγματικα εκπλησουμε Επιτροπή να υποβάλει παρατηρήσεις όσον αφορά τα δικρώμενα συμφέροντα χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά προβλήματα νομικά όσον αφορά τα δικαιώματά τους στον Καναδά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταφορά αρμοδιοτήτων και τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων των ευρωπαϊκών στην αγορά του Καναδά αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να προστατευθούν με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Παίρνω το λόγο με την ιδιότητά μου του συντονιστή της ομάδας ΕΝΕΛ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλά υπόθεση, στην Επιτροπή μάλλον αυτήν εδώ. Ε, πολλά έχουν υποθεί για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να πω ότι η συνθήκη αυτή, όπως ο μεγάλος της αδελφός, η η TTIP συντάχθηκε ε, στο πλήρες σκοτάδι. Να σχολιάσω το πρόβλημα στο γεωργικό τομέα, γιατί σήμερα λαμβάνει χώρα η γεωργική σύνοδος εδώ στη Βρυξέλλες και οι γεωργοί, οι αγρότες θα πληγούν ιδιαίτερως από τη συμφωνία με τον Καναδά, κυρίως οι κτηνοτρόφοι, οι εκτροφείς ε, χοιρινού και βοδινού, ε, παραγωγή χοιρινού και βοδινού κρέατος. Είδαμε εδώ ότι θα υπάρξουν δικαιοδοτικά όργανα, διαιτητικά, τα οποία θα δώσουν δίκαιο πάντοτε στις πολυεθνικές σε των ε, κρατών. Πριν από λίγες μέρες συμμετείχα σε μια ομάδα εργασίας για τη Συμφωνία ΣΥΤΑ και με λίγο μου διαπίστωσα ότι για άλλη μια φορά μόνο 140 ε, ΠΟΠ θα προστατευτούν, ενώ σήμερα έχουμε χιλιάδες ΠΟΠΟ, προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευση και απειλούνται όλα αυτά στην Ευρώπη. Αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ΣΥΤΑ είναι μία ε, ανταλλαγή συναλλαγών αλλά δεν πρέπει να το αναμίξουμε με το TTIP, γιατί θα κάνουμε ολέθριο σφάλμα. Πρόκειται, εν πάση περιπτώσει, για μία πρώτη συμφωνία μεταξύ των δύο πιο βιομηχανοποιημένων περιφερειών. Μπορούμε να πιστεύουμε σε αυτό, αλλά για πρώτη φορά μία διεθνής ε, σύμβαση επιτρέπει στους επενδυτές να ε, παραπέμψουν στα δικαστήρια τους ε, δικούς μας φορείς γιατί αυτό μπορεί να αφορά από τις ορμόνες στο κρέας μέχρι τα πετρελαϊκά υποπροϊόντα. Δηλαδή τι κάνουμε, βραχικυκλώνουμε τις ε, διεθνείς συμβάσεις όταν θέλουμε μία αδρή αποζημίωση και αυτό αφορά ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο θα στοιχήσει 400.000 ε, ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεχνάμε την εθνική κυριαρχία. Όπως ε, ελέγχθη πρόσφατα, δεν μιλάμε για δικαιώματα μόνο των Καναδών επενδυτών, αλλά και εκείνων που έχουν θρηγατρικές και στην Ευρώπη. Μιλάμε για 47.000 επιχειρήσεις αμερικανικές που θα είχαν πρόσβαση μέσω TTIP στο ίδιο δικαστήριο. Ε, παρά τις ε, εγγυήσει της Επιτροπής δεν νομίζω ότι το θέμα της διατροφικής ασφάλειας έχει λυθεί. Το θέμα των ορμονών υπάρχει και θα πρέπει να εξευρεθεί ένας μηχανισμός έτσι ώστε να αποφευθούν οι κίνδυνοι. Θα πρέπει λοιπόν ε, τα ε, γενετικώς τρεποποιημένοι οργανισμοί να την χάνουν ελέγχου, ιδιαίτερα σε σχέση με το κρέας. Τέλος, το ΣΥΤΑ ε, δέχεται τις 145 γεωγραφικές ενδείξεις από τις χιλιάδες. Και ξεχνάμε τους μικρούς επιχειρηματίες. Εγώ δεν αντιτάσσομαι στο εμπόριο. Γιατί χρησιμοποιείται όμως οι ελεύθεροι, γιατί χρησιμοποιούνται οι ελεύθερες συναλλαγές για να μην λαμβάνουμε υπόψη το διεθνές εμπόριο Τζουντ. Πολλά ελέγχθησαν, υπάρχουν καλά και αρνητικά στοιχεία τα οποία θα αποτιμήσουμε πριν από την έγκρισή μας. Η Επιτροπή είπε ότι δεν θα ξανανοίξουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά το αδύνατο πολλές φορές γίνεται δυνατό. Το είδαμε ήδη αυτό. Καταρχήν το Συμβούλιο από τις τελευταίες ε, διαπραγματεύσεις ασχολείται με τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότησή τους. Αυτή είναι η πρώτη εμπορική συμφωνία με βάση ένα αρνητικό κατάλογο. Γιατί δεν λαμβάνουμε αυτό το βαθμολόγιο με βάση την πρόταση για την επίλυση διαφορών γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης προστασία όπως είπατε. Το δεύτερο που αφορά την επίλυση διαφορών επενδυτή κράτους. Ξέρετε ότι τον Ιούλιο με βάση το TTIP είπαμε ότι θα πρέπει να ε, σεβαστείτε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πώς ε, τηρείται αυτό, αυτή η προδιαγραφή με βάση τη νέα ΣΥΤΑ όπως ορίζεται. Μαρία. Θα ήθελα να παρέμβω πολύ πιο συγκεκριμένα πώς ξέρουμε πώς ορίζεται η επίλυση διαφορών, πώς δηλαδή οι Καναδοί ζητάνε να προστατευτούν έναντι των ε, διαφορών με τους Ευρωπαίους επενδυτές. Ξέρουμε ποιος θα καλύψει τα έξοδα αυτού του Διεθνούς Δικαστηρίου. Έχουμε ορίσει τη σχέση ε, που υπάρχει με βάση μια καλύτερη ρύθμιση, better regulation, πώς θα βελτιώσει τις επενδύσεις. Τι νόημα έχει να υπάρχει ένας μηχανισμός επίλυσης διαφόρων. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ο Καναδάς είναι απομονωμένος. Εσείς μιλήσατε πρόσβαση για την πρόσβαση στις αγορές. Μιλήσαμε για μια συμφωνία, την συμφωνία Τίζα, σε σχέση με τις υπηρεσίες. Υπάρχει και ένας ε, θετικός κατάλογος. Δεν υπάρχει στον ΠΟΕ. Γιατί επιλέξατε έναν θετικό κατάλογο. Επίσης, οι Γερμανοί στις επιφυλάξεις μίλησαν και για τις υπηρεσίες υγείας. Οι Γερμανοί ανησυχούν για τις υπηρεσίες αυτές ή υπάρχει πραγματικά κίνδυνος. Είπατε ότι θα γίνουν διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο. Ε, δεν ξέρω αν κατανόησα καλά. Αυτό που μας απασχολεί είναι η κύρωση. Δηλαδή θα μπορούσε να τεθεί ενισχύ αυτή η συμφωνία χωρίς την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπούχνερ. Ευχαριστώ πολύ το Γενικό Διευθυντή για τα πολύ θετικά σχόλια που έκανε και την πολύ θετική παρουσίαση. Πολλοί οργανισμοί αλλά και εμπειρογνώμονες για θέματα εμπορίου έχουν εκφραστεί πολύ επικριτικά και τελικά βλέπουμε ότι και η νομική βάση αλλά και από την άποψη του χρήστη και των επιχειρήσεων έχουν εκφράσει επικρίσεις. Υπάρχει επίσης, όπως ξέρετε, και η πολύ συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη από μέρους των Γερμανών δικαστών οι οποίοι εκφράστηκαν κατά αυτού του συστήματος επίλυσης των διαφορών και αναρωτιέμαι πραγματικά αν εσείς θεωρείτε ότι όλοι αυτοί, από όπου και αν προέρχονται οι κριτικές, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εκφράστηκαν κατά έχουν ε, εσφαλμένη άποψη και αν είναι σωστό να επιλέξουμε παρόλα αυτά αυτά τα ε, συστήματα επίλυσης των διαφορών τα οποία δεν έχουν την εγγύηση αν θέλετε του ε, πραγματικού δικαστή. Θα ήθελα να αναγνωρίσουμε ότι εδώ υπάρχει τουλάχιστον αμφισβητούμενη προσέγγιση και όσον αφορά τις εισαγωγές βόλιου και χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε και εδώ πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Εξάλλου στο έγγραφο που μας προτείνεται υπάρχουν και άλλες προτάσεις οι οποίες μου φαίνεται ότι είναι πολύ πραγματοποίηση. Κύριε Ντεμαρτή, λέει κυρία Λεπέν, πρόκειται για μια πρόταση η οποία βλέπουμε να εμφανίζεται, να εξαφανίζεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανάλογα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους σας. Εδώ και 1,5 χρόνο έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και έχω την εντύπωση ότι περιμένετε με ποιο τρόπο θα το περάσετε χωρίς να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τι ακριβώς κάνετε. Είστε ένας γραφειοκράτης, δεν είστε εκλεγμένος και δεν εκπροσωπείτε κανέναν λαό της Ευρώπης. Καλό θα ήταν αν δείχνατε λίγο ε, θάρρος να μην κρυβόσαστε πίσω από όλα αυτά τα σύγχρονα κτίρια των ευρωπαϊκών κτίριων. Βλέπουμε ότι το κόστος ε, των κτηνοτρόφων της ε, Αμερικής αλλά και του Καναδά είναι κατά 30% χαμηλότερο από αυτό των Ευρωπαίων ε, γεωργών και κτηνοτρόφων. Θα καταφέρετε λοιπόν να τους εξοντώσετε. Βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά θα αποτελέσετε αυτές ε, τις αρχές οι οποίες ε, δίνουν ένα πολύ θανατηφόρο χτύπημα στους Ευρωπαίους οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία όταν υπάρχουν διαφορές, αυτές θα προβλέπει ότι όταν υπάρχουν διαφορές αυτές θα επιλύονται από ένα όργανο το οποίο βρίσκεται εκτός της Ευρώπης, πρόκειται για ένα ιδιωτικού δικαίου και παρά τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν εδώ και 1,5 χρόνο, από ό,τι διαπιστώνω, οι πρόσφατες αλλαγές είναι καθαρά καλοπιστικές. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν επιλύονται τα προβλήματα τα και οι δυσκολίες οι οποίες έχουν ε, εντοπιστεί από Ευρωπαίους αλλά και άλλους ε, επικριτές. Και αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, το κείμενο για την αντίρρηση όσον αφορά την επίλυση των διαφορών και το Διαιτητικό Δικαστήριο έχει υπογραφεί από πάνω από 3,5 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Θα τους αγνοήσετε. Για άλλη μια φορά δείχνετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα αυταρχικό τοταλιστερό πρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να εξετάσουμε τη συμφωνία κεφάλαιο προς κεφάλαιο, το καθένα ξεχωριστά και να διαβάσουμε πολύ προσεκτικά τι περιέχεται στο κείμενο, έτσι ώστε να έχει ο καθένας και κάθε μία από εμά την πλήρη ενημέρωση για το περιεχόμενο του κειμένου. Γιατί δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι όλοι έχουν διαβάσει τις 1600 σελίδες και έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο του εγχειρήματος. Ζωλίκ, ε, μπορείτε να έχετε το λόγο για να απαντήσετε και κυρίως να μας μιλήσετε για το χρονοδιάγραμμα. Ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα, ε, ποια, ε, ποιες είναι οι ημερομηνίε κλειδιά για την συνέχεια που θα δοθεί στη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας. Ο Ζωλίκ, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ως προς το χρονοδιάγραμμα. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. πότε θα ολοκληρωθεί η μετάφραση του κειμένου των 1600 σελίδων. Να σας υπενθυμίσω ότι εργαζόμαστε πάνω σε 23 γλώσσες και οι γλωσσικές και μεταφραστικές υπηρεσίες είναι αρκετά γρήγορες, ωστόσο χρειάζεται χρόνος και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να υποβάλει το κείμενο αυτό προς υπογραφή τον Ιούνιο και να διαβεβαιώσω ότι κυρία Σάκε δεν μπορεί κανείς να πάει πιο γρήγορα. Προχωρούμε εξαιρετικά γρήγορα. Σαφέστατα υπάρχει κόστος και τιμή στη δημοκρατία και οφείλουμε να αναλάβουμε αυτό το τίμημα και αυτό το κόστος και γι' αυτό το σύστημα μας είναι ε, μακροσκελές γιατί είναι πολύ δημοκρατικό και διαφανές δεν μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα. Γι' αυτό και το κείμενο θα είναι έτοιμο προς υπογραφή τον Ιούνιο. Θα υποβληθεί στο Συμβούλιο ε, ε, τον Ιούνιο προς υπογραφή και τον Οκτώβριο μάλλον θα έχουμε διμερή σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά όπου θα υπογραφεί επισήμως και μετά θα υπάρχει συγκατάθεση, consent στα αγγλικά και ratification, κύρωση ε, στα γαλλικά, όχι διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ε, ε, ο Κάριλ Ντεγκούρτς, ο πρώην Επίτροπος, στην ακρόασή του το 2009 είχε πει ότι δεν μπορεί να υπάρχει προσωρινή εφαρμογή πριν από την κύρωση, ratification, από, την, αυτό το κοινοβούλιο. Συγκατάθεση, δηλαδή consent. Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως δεν θα υπάρχει προσωρινή κύρωση στο βαθμό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Και για τα εθνικά κοινοβούλια είναι η ερώτηση. Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, λέει ο Ζων Λουίκ. Εάν πρόκειται για μεικτή συμφωνία και προς το παρόν η Επιτροπή ε, θα επιφυλάσσεται να απαντήσει, το Συμβούλιο θεωρεί ότι πρόκειται για μεικτή συμφωνία. Δεν υπάρχει παράδειγμα συμφωνίας που αποφασίστηκε ως ε, ούσα μεικτή συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση Η προσωρινή εφαρμογή λαμβάνει χώρα μόνο στο σκέλος που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από κοινού αρμοδιότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτους μέλους εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητά της. Δηλαδή η τελική κύρωση του κειμένου θα έχει ολοκληρωθεί ε, εάν όταν θα το έχει κυρώσει κάθε εθνικό κοινοβούλιο και μάλιστα και περιφερειακό κοινοβούλιο, π.χ. στην περίπτωση του Βελγίου. Και ο... μέχρι ότου ολοκληρωθεί αυτό, δεν θα έχει υπάρξει επίσημη ε, κύρωση πλήρως της συμφωνίας. Εγώ, εμένα μου αρέσει να μιλάω για τα γεγονότα και θα προχωρήσουμε με βάση τις προηγούμενες συμφωνίες με την ε, Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προχωρήσουν τον τρόπο που έχουν προχωρήσει και στο παρελθόν. Μπορώ να συνεχίσω. λέγοντας ότι είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία και νομίζω ότι αξίζει να χάσουμε λίγο χρόνο, να εξοδεύσουμε λίγο παραπάνω χρόνο για αυτή, να μην αφήσω ερωτήματα αναπάντητα για τα θετικά σχόλια του κυρίου Πάμπριξ. Πράγματι, συμφωνούμε, έτσι βλέπουμε και εμείς τα πράγματα. Το μάντρα που μας χαρακτηρίζει, δηλαδή το σλόγγαν, το σύνθημα που μας ε, ε, χαρακτηρίζει είναι υποσχόμαστε λιγότερα και τελικά παραδίδουμε και προσφέρουμε, ε, εκπληρώνουμε περισσότερα. Είναι αυτή η βασική αρχή που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε με πλήρη μετριοπάθεια. Τώρα, ως προς τα διάφορα ερωτήματα για το σύστημα το δικαστικό για την επιλύση των συγκρούσεων σε θέματα επενδύσεων, για τη διαιτησία, για το ότι δεν είναι δημοκρατικό το σύστημα αυτό. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι είμαστε μπροστά σε ένα νέο μοντέλο προστασία του δικαιώματος του νομοθετήν, του νομοθετήν ανεξάρτητο μόνιμο δι, δικαστήριο πρώτο βάθμιο και το ίδιο για, το, για τις εφέσεις, για την δευτεροβάθμια εκδίκαση των υποθέσεων. Είναι η αρχή ε, τριών ε, κλειδιών, αν θέλετε. Ε, τρεις βασικές αρχές κλειδιά. Αυτό αντιτίθεται με το παρελθόν σύστημα του ISDS, του Διεθνούς Συστήματος για την Επίλυση των Συγκρούσεων. Οι, κάποιοι δικαστές, οι δικηγόροι του ISDS, δεν τους αρέσει ιδιαίτερος αυτού, αυτό που κάνουμε, ενδεχομένως γιατί μειώνεται έτσι το κομμάτι της πίτας που θα υπάρχει για αυτούς. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τι ακριβώς κάνουμε. Σε πάρα πολλά συστήματα Υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης στην ε, εγχώρια νομοθεσία. Δεν ισχύει αυτό στην Ευρώπη. Όμως στη είπα, ή στο Καναδά μπορεί κανείς να κάνει αυτή τη διαφοροποίηση στην εγχώρια νομοθεσία και αυτό το έχουν αποδείξει στο παρελθόν. Δεύτερον, οι συμφωνίες αυτές δεν είναι άμεσα εφαρμόσεμες και αν δεν υπάρχει ένα σύστημα επίλυσης διαφορών και γι' αυτό υπάρχει άλλωστε ένα τέτοιο σύστημα σε όλες τις συμφωνίες, όχι μόνο τις επενδυτικές αλλά και τις άλλες, θα μπορούν οι επενδυτές ενδεχομένως να διατρέχουν το κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις από τα εγχώρια δικαστήρια στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά ή αλλού στον κόσμο γιατί δεν θα τη χάνουν προστασίας από τη συμφωνία η οποία δεν θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη. Αυτή είναι η βασική αιτία, είναι ένα βασικό στοιχείο. Στόχος μας είναι να έχουμε ένα επίπεδο προστασίας για τους επενδυτές μας στο εξωτερικό που να είναι κοντά στο επίπεδο προστασίας που έχουν οι επενδυτές μας στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση τα πρότυπα ε, είναι κάπως χαμηλότερα από τα δικά μας ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει περισσότερη προστασία από ό,τι στο δικό μας σύστημα, αλλά κάπως λιγότερη. Αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να τους προστατεύσουμε ούτως ή άλλως. Και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να προστατεύσουμε και τους επενδυτές της τρίτης χώρας. Και είναι σαφές ότι οι επενδυτές της τρίτης χώρας συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα να ε, προσφύγουν στα δικά τους εγχώρια δικαστήρια αν θεωρούν ότι τα πρότυπα εκεί είναι καλύτερα. Και δεν υπάρχει καμία σύγχυση, γιατί εάν ένας επενδυτής προσφύγει στα εγχώρια δικαστήρια, δεν μπορεί να προσφύγει στο μηχανισμό διαιτησίας για την επίλυση ε, των συγκρούσεων. Θα πρέπει ο επενδυτής κάποια στιγμή να διαλέξει, δεν μπορεί να κάνει και τα δύο. Αλλά ε, δεν είναι ο βέλτιστος, δεν είναι τέλειος ο κόσμος μας, αλλά προσπαθούμε να έχουμε το βέλτιστο δυνατό είναι μια, σαφής, μια σαφή επιλογή την οποία θα πρέπει να κάνουν οι επενδυτέ. Είναι βασικό στοιχείο αυτό, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και ε, πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο. Τώρα, ως προς τη γνώμη των ε, Γερμανών δικαστών που αναφέρθηκε, αυτό το οποίο με εκπλήσει είναι ότι για 50 χρόνια είχαμε στο παρελθόν 1 ή 100 και διμερείς συμφωνίες ε, το 95% χωρίς ιδέες ή με πεπεβαλαιωμένες ιδέες, το υπόλοιπο 5% με ιδέες ή πιο φρέσκες ιδέες και για όλες αυτές τις 100 και διμερείς συμφωνίες μεταξύ γερμανικής ε, μεταξύ Γερμανίας και άλλων χωρών οι Γερμανοί δικαστές ποτέ ε, δεν αναρωτήθηκαν ή δεν τις αμφισβήτησαν ή δεν τις ε, απόρριψαν και αυτό με προβληματίζει κάπως. Έτσι έχει η κατάσταση, νομίζω ότι σας απάντησα. Και αν θέλουμε να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τους επενδυτές μας έναντι των διακρίσεων που υφίστανται στο εξωτερικό, θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα όπου ε, να παρέχουμε προστασία γενικότερη, με δημοκρατικό τρόπο να ορίζονται οι αρχές, οι δικαστικές, σίγουρα πρόκειται για μια νέα προσέγγιση και τη χρησιμοποιούμε σε όλες μας τις διαπραγματεύσεις και με την TTIP και στο πλαίσιο της TTIP και δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα το πετύχουμε αυτό με τους Αμερικανούς. Αν όμως δεν το πετύχουμε με τους Αμερικανούς είναι πολύ απλά τα πράγματα, δεν είμαστε έτοιμοι να ε, συμβιβαστούμε και να επαναχωρήσουμε έναντι των τριών βασικών αρχών που ανέφερα προηγουμένως. Σε όλες τις διαπραγματεύσεις μπορεί να υπάρχουν κάποιες προσαρμογές, αλλά οι προσαρμογές αυτές δεν μπορούν να αλλοιώνουν τα στοιχεία κλειδιά, τις αρχές κλειδιά ε, που ε, αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος προς αυτό. Για τις επενδύσεις λοιπόν νομίζω ότι κάλυψα, απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Έρχομαι τώρα στις λοιπές ερωτήσεις και θα μιλήσω γαλλικά για το θέμα της γεωργίας. Επομένως, για τη γεωργία να πω τα εξής. Να σας υπενθυμίσω τους στόχους που επιδιώξαμε. Με τον Καναδά το εμπόριο είναι κάπως ε, ε, πλέον ασματικό ως προς τα διατροφικά προϊόντα, τα προϊόντα σύντησης και τη γεωργία γενικότερα. Έχουμε πολλά επιθετικά συμφέροντα στη δική τους αγορά, κυρίως στο γαλακτοκομικό τομέα, 20.000 ε, τόνους τυριού μας έχουν δώσει πάρα πολύ καλούς δασμούς να το πω. Αυτό που μας προσφέρουν οικονομικά στις δικές μας ε, επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επομένως στο γαλακτοκομικό τομέα κερδίζουμε αρκετά. Τώρα, ως προς τους εκτροφείς, οι 46.000 τόνοι που ανέφερε ο συνάδελφος είναι το μισό της εκατό της αγοράς μας και θα έχουμε 0,3% ε, της αγοράς μας. 0,5 και 0,3 λοιπόν θα είναι το απόθεμα αντίστοιχα στο χοιρινό και στο βοδινό κρέας. Ε, και όντως ε, τα κτηνοτροφικά είναι ο τομέας στον οποίο θα έχουμε εμεί αμυντική στάση εναντί των Καναδών, ενώ στο γαλακτοκομικό έχουμε επιθετική στάση εναντί των, Καναδών. Και θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να μην αποσταθεροποιηθεί ο τομέας της κτηνοτροφίας με την Ιαπωνία και την Κορέα είμαστε άμεσα ανταγωνιστικές χώρες ή υπάρχουν χώρες πολύ πιο ανταγωνιστικές από ό,τι είμαστε ε, εμείς. Ποτέ δεν θα απελευθερώσουμε πλήρως την αγορά των πουλερικών του χοιρινού του βοδινού κρέατος ως προς τις χώρες αυτές που είναι απολύτως ανταγωνιστικές έναντι ημών. Όμως ο Καναδάς δεν είναι και γι' αυτό μπορούμε να το απελευθερώσουμε μερικώς αυτή την αγορά, κερδίζοντας κάπου αλλού βέβαια. Έχουμε μια συμφωνία για το κρασί με τον Καναδά που προστατεύει εκατοντάδες ε, προστατευόμενες ονομασίες προέλευση. Έχουμε 145 ε, δείξεις γεωγραφικές που θεωρήθηκαν προτεραιότητα από τα κράτη-μέλη και γι' αυτό θα τις προστατεύσουμε όλες το ίδιο με λίγες εξαιρέσεις που υπάρχουν και στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόλου δεν απειλούνται οι ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης, αλλά αντίθετα έχουν προστιθέμενη αξία. Και στο μέλλον, για παράδειγμα, το προσούτο της Πάρμας μπορεί να τίθεται σε εμπορία στον Καναδά, ενώ δεν μπορούσε μέχρι σήμερα. Διότι υπάρχει trademark, υπάρχει εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα Πάρμα στο Καναδά και δεν είχε με τέτοιο δικαίωμα. Επομένως, πολύ καλή προστασία και πολύ καλό αποτέλεσμα και για τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης. Ως προς... Να δω τις σημειώσεις μου για το χρονοδιάγραμμα απάντησε, για τη Γεωργία επίσης και τις προθεσμίες. Ως προς τα ερωτήματα του κυρίου Ζαντό να πω ότι δεν διαπραγματευόμαστε τους κανονισμούς μας. Αναφερθήκατε στον κανονισμό για την ποιότητα των καυσίμων, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, ο κανονισμός αυτός δεν αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης με τον Καναδά. Ποτέ δεν είχαμε την πρόθεση και δεν έχουμε την πρόθεση να διαπραγματευτούμε τους δικούς μας ευρωπαϊκούς κανονισμούς με τον Καναδά. Αναφερθήκατε στη μελέτη του κυρίου Μέσελεν για τις δημόσιες αγορές και αυτό το δείχνει ότι το άνοιγμα των δημόσιων αγορών στη ΣΥΠΑ και στο Καναδά θα είναι, με τι θα είναι συγκρίσιμο αναρωτιέστε. Ουσιαστικά σε αυτή τη μελέτη αναφέρεστε έχω την εντύπωση και η μελέτη αυτή έχει ένα μεγάλο σφάλμα. Δεν αναφέρεται παρά μόνο σε ένα μικρό μέρος των τρόπων με τους οποίους οι δημόσιες αγορές ανοίγουν για τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών, στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Δηλαδή, Μιλούμε για τις διασυνοριακές ε, δημόσιες αγορές όπου επιχειρήσεις στις τρίτες χώρες παίρνουν συμβόλαια ε, στην γειτονική χώρα. Αυτό αντιστοιχεί στο 4% των, ε, της συνολικής αγοράς, του συνόλου των δημοσίων αγορών και η μελέτη έχει αυτό το σφάλμα, αυτή την έλλειψη. Με θηγατρικές και με συμμετοχή σε κοινοπραξίες το μπορούν οι επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στις δημόσιες αγορές και μάλιστα σε ένα ποσοστό πενταπλάσιο ή τετραπλάσιο του 4% και μάλιστα ε, το νούμερο του 4% υπάρχει στην, για την Ευρώπη. Στη ΣΥΠΑ δεν έχει γίνει τέτοια μελέτη. Η αγορά των ΗΠΑ ήταν πολύ πιο κλειστή από ότι η ευρωπαϊκή και αυτό θέλουμε να καμφθεί στη διαπραγμάτευση TTIP και αν δεν τα καταφέρουμε γι' αυτό έχουμε και τροποποιημένη πρόταση για το εργαλείο αμεβαιότητας στο θέμα των δημοσίων αγορών και ότι στόχος μας είναι οι επιχειρήσεις να μπορούν να συμμετάσχουν σε περισσότερες δημόσιες αγορές. Τώρα ως προς τον αρνητικό κατάλογο, negative list, που αναφέρθηκε για τον τομέα των υπηρεσιών, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο αρνητικός κατάλογος είναι ένα εργαλείο μόνο. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι το αποτέλεσμα και θα συνεχίσουμε όπως το κάναμε και στο παρελθόν να προστατεύουμε τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες προστατεύονται σε αυτή τη συμφωνία όπως προστατεύονται και σε όλες μας τις συμφωνίες. Και αυτό τι σημαίνει. Και σας υπενθυμίζω. για την υγεία, για την εκπαίδευση, για τις κοινωνικές υπηρεσίες, για τη διανομή του νερού. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Είμαστε απολύτως ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι επιθυμούμε. Και Συν της άλλης υπάρχουν και οι υπηρεσίε κοινή ωφέλεια. Η επιφύλαξη δηλαδή που έχουμε για ε, κοινή ωφέλεια και υπηρεσίε κοινή ωφέλεια και εκεί έχουμε το ελεύθερο να έχουμε το μονοπόλιο που επιθυμούμε ως προς την πρόσβαση στην αγορά για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ε, θα θέλαμε να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε. Η μόνη υποχρέωση για αυτό το σκέλος που δεν έχει να κάνει με την υγεία, που δεν έχει να κάνει με το νερό, που δεν έχει να κάνει με την κοινωνική υπηρεσία, ε, τις κοινωνικές υπηρεσίες και το καθεξής, Εάν κάτι είναι ανοιχτό προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, τότε να μην υπάρχουν διακρίσεις. Αυτή είναι η μόνη μας υποχρέωση και ο μόνος περιορισμός. Αν κάτι ήδη έχει απελευθερωθεί και, και μπορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση, ε, τότε να γίνεται χωρίς διάκριση έναντι των επιχειρήσεων. Μεταξύ τους μάλλον. Είναι σαφές και θα συνεχίσουμε το πράττουμε και στο ε, μέλλον. Στο παρελθόν κανείς ποτέ δεν έχει Κανείς ποτέ δεν, έχει, ε, δεν το έχει αυτό αφισβητήσει. Τώρα, νομίζω ότι απάντησα στα περισσότερα ερωτήματα. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις εναντί των σχολείων της κυρίας Λεπέν. Ναι, είμαι αξιομετούχος σε ψηλή ε, θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαι Γάλλος και είμαι περήφανος γι' αυτό. Δεν είμαι ερετός και δεν πρόκειται να διεκδικήσω ερετή θέση, αλλά είμαι ε, διατεθειμένος να συζητήσω με τον οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε φόρουμ, σε οποιοδήποτε βήμα και σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης έχω ε, τη συνήθεια και έχω εκπαιδευτεί να κάνω διάλογο με πολύ δύσκολους συνομιλητές και σε πολύ δύσκολα φόρουμ. Μην ανησυχείτε καθόλου. Εμείς λειτουργούμε στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, έτσι όπως το κάναμε μέχρι και σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να αποφανθεί και αν τελικά η συμφωνία αυτή θεωρηθεί μεικτή συμφωνία θα αποφανθούν και τα ε, εθνικά κοινοβούλιο. Μπορεί ε, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν ταχθεί κατά αυτής της συμφωνίας στο διαδίκτυο μέσω συγκέντρωσης υπογραφών, το σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο εκπροσωπούνται στα εθνικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για το ΣΥΤΑ όταν μεταφραστεί το κείμενο. Τον Ιούνιο λοιπόν η ίντα θα αρχίσει με συγκεκριμένη εργασία επί του κειμένου. Ευχαριστούμε πολύ Ζαν Λουκ για αυτή την εισήγηση και τώρα κλείνει η συνεδρίαση για το κοινό και θα συνεχίσουμε και κλεισμένων των θυρών. Άρα μόνο οι βουλευτές, πολιτικές ομάδες, βοηθοί και γραμματεία μπορούν να παραμείνουν. Θα ήθελα οι φιλοξενούμενοι μας, οι ακροατές μας να